δήλωση ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία του είδους αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ε, πρόκειται για πολυπληθείς ψηφοφορίες. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και βάσει της απλουστευμένης διαδικασία ε, πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση τη κυρίας Παλιαδέλη σχετικά με το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστική Κληρονομιά. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορία. ψήφισαν 556 υπέρ 497 κατά 18 41 αποχές συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πρέπει τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία της κυρίας Πάκα σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Νομοσπονδίας στο πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση και στο πρόγραμμα Δράση του τομέα της μάθησης διαβίου. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Σάιερ σχετικά με τον έλεγχο από πλευρά κρατών μελών της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Εξετάζουμε λοιπόν την πρόταση. Έχουμε 25 τροπολογίες νομικής επιτροπής. Ψηφίζουμε unblock, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, πάντα κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 28 στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 καταπίπτει. Μετά το, την Παύλα 14, τροπολογία 31 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα για το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ολοκληρώθηκε. 589 ψηφίσαντες, 567 υπέρ, 4 αποχές, 18 αποχές και επομένως εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Αντρικιενέ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Εξετάζουμε λοιπόν την πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 245 ψήφοι υπέρ, 348 κατά, μία αποχή, επομένως η τροπολογία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 11, πάλι διονομαστική κλήσεως. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 302 ψήφοι υπέρ, 282 κατά 9 αποχές, επομένως η τροπολογία εγκρίνεται. Παράγραφος 54, ε, τροπολογία Howitt. Όχι, λέει η Πρόεδρος. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία 12, διονομαστικής ε, ψηφοφορίας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. «138 ψήφοι υπέρ, 457 κατά, 138 ψήφοι υπέρ, 457 κατά. Όχι. Κύριε Σιλβέστρης, πέστε μας. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που προσπαθούν να πούν κάποιοι συνάδελφοι είναι ότι μπορείτε να λέτε ότι εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε χωρίς να λέτε τόσοι υπέρ, τόσοι ψηφίφαντες κτλ. Ναι, ε, σα είπα απλώ τι φώναζαν οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Ε, ωραία, η τροπολογία λοιπόν 12 έχει απορριφθεί. Ε, προφορική τροπολογία Χάουιτ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Είναι ένα θέμα ουσία. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αφαιρθούν λέξει στην Κροατία. Νομίζω ότι δεν είναι αμφιλεγόμενο με τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Υπάρχουν αντιρρήσει. Εντάξει, επομένως μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, προφορική τροπολογία του κυρίου Χάουιτ επί της παραγράφου 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 2 και 5 που είναι ταυτόσιμες. Δύο ονομαστικής ε, ψηφοφορίας. Παρακαλώ, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 83 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία το, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία αυτή απερίφθη. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στο δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας και της επόμενης εμείς έχουμε ζητήσει, η ομάδα μας θα ακολουθήσει ελευθερία ψήφου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 25 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Η παράγραφος 115 καταπίπτει επομένως. Ψηφίζουμε την τροπολογία 13 ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 14 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία 14 απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 15, πάντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Έχουμε τώρα δύο προφορικές τροπολογίες των Λοχ Μπίλερ και Αντρίκινε. Επί της τροπολογίας 7 θέλετε το λόγο. Υπάρχουν δύο προσθήκες στο κείμενο, λέει. Ο κατάλογος των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η ε, βιασμοί, ε, λογοκρισία και στην περίπτωση του Ιράν λέμε εξοδικαστικές εκτελέσεις. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Περνάμε τώρα λοιπόν στην προφορική τροπολογία της κυρίας Αντρίκενε. Κυρία Αντρίκενε, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε και εμεί μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7. Το κείμενο θα λέει τα εξή. Ζητά από την Κομισιόν να καταρτήσει ένα κατάλογο ατόμων που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπω βασανιστήρια, βιασμοί, ε, λογοκρισία και, εξοδικα... και εκτελέσεις στο Ιράν, ιδίω μετά από τι εκλογέ του 2009 και να εξετάσει η Κομισιόν τη δυνατότητα να υπάρξει, υπάρξουν κυρώσεις με, την, με το πάγμα των στοιχείων του ενεργητικού τους και απαγορεύσει ταξιδιού. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν. Συμφωνούμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 140. Επ' αυτή σε προτείνει προφορική τροπολογία η κυρία Αντρίκεν. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις στην Ρωσία. Επομένως, θα θέλαμε να αλλάξουμε την φράση που αρχίζει και λέει ότι ε, δυστυχώς ε, όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει προσέκρουσαν στην άρνηση των αρχών. Άρα να αντικαταστήσουμε τις λέξεις so far στον αγγλικό μέχρι τώρα ε, με το να πούμε, ε, για να πούμε μέχρι 31 ε, Οκτωβρίου 2010. Κάνεις αντίρρηση. Όχι, επομένω ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 140 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 9 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 17. Συγγνώμη, την τροπολογία 16 πρώτα, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 17, διανομαστικής ψηφοφορίας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ε, στην εισηγήτρια. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση Αρλάκη, μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Περνάμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίζουμε πρώτα την παράγραφο 2 ε, σε χωριστά τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίθηκε. Παράγραφος 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 και έχουμε μία προφορική τροπολογία Κιλ Νίλσεν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μία τροποποίηση της πρώτης λέξης της τελευταίας φράσης της παραγράφου 30 να αντικαταστήσουμε το χαιρετίζει με το καταγράφει. Ci sono Αντίθετες απόψεις, όχι. Επομένως ε, ψηφίζουμε την παράγραφο 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 37 κατά τμήματα ε, και με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Παράγραφο 40, κατά τμήματα, τρία τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 44 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη η τροπολογία. Παράγραφος 52. Κατά τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 56. Κατά τμήματα και έμενο μας και η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 66. Προφορική τροπολογία Αρλάκη. Παρακαλώ. Μετά από συζητήσεις με άλλες πολιτικές ομάδες προτείνω να αλλάξει ε, η παράγραφος 66 και να λέει «Σημειώνει ότι η ανάμειξη των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν ε, έτσι και να διαβεβαιώσουμε ότι το Πακιστάν ε, θα έχει ικανοποιητική λειτουργία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Non 40 Δεν βλέπω να είναι 40 οι βουλευτές που αντιτίθενται. Επομένως θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία υπέρ κατά ονομαστική, ονομαστική, ονομαστική ψηφοφορία. Δεν μέτρησα 40 βουλευτές, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Α, όχι, λέει η Πρόεδρος, ονομαστική ψηφοφορία, εντάξει. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Παράγραφος 67 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Παράγραφος 71. Τροπολογία προφορική του κυρίου Αρλάκη στο τρίτο τμήμα του κειμένου. Παρακαλώ, προτείνω να αλλάξουμε ολόκληρο το, το τμήμα 3 της παραγράφου 71, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι ειδικέ δυνάμεις και η τοπική αστυνομία ε, θα προχωρήσει σε δράση κατά των Ταλιμπάν έχοντας πλέον μηδενική ανοχή προς ε, ε, πράξεις εναντίον των αμάχων. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επομένως ψηφίζουμε την παράγραφο 71 με τέσσερα σε τέσσερα τμήματα. Ξεκινούμε πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Η ομάδα Άλτε προτείνει το τέταρτο τμήμα της παραγράφου 71 να γίνει μια ξεχωριστη παραγραφο παράγραφος 71α. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, επομένω ψηφίζουμε την παράγραφο 72 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 73 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέρας. Εγκρίνεται. 81 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραφρός 88 πάλι με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Παράγραφος 89 κατά τμήματα με ονομαστική κλίση πρώτο τμήμα και πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται παράγραφος 93 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G, λατινικό, κατά τμήματα και μονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θεολογική σκέψη M, λατινική. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. ακολουθεί το ψήφισμα τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για τη δημιουργία ενό μόνιμου μηχανισμού διαχείριση των κρίσεων και για την διατήρηση τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Τροπολογία 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχε. εγκρίνεται. Παράγραφο 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, μια στιγμή. Ο κύριος Σάντζεφ Πεσέδο θέλει να κάνει μια τεχνική διευκρίνηση. Όχι. Ναι κύριε Πρόεδρε ως ε, συντάκτης της τροπολογίας υπαριθμών 9 εκεί που λέει M-E-E θα πρέπει να λέμε e κάθετος e Ευχαριστώ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Έχει αποσυρθεί. Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 9 κατά τμήματα, δύο τμήματα, με ονομαστική κλίση, πρώτο τμήμα. Απλή ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10, τροπολογία 10, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 6, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Hughes έχει προτείνει μια προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 12. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Σοσιαλιστέ Δημοκράτε, το ΕΛ και οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι κατεβάζουμε αυτή την τροπολογία και απευθύνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόσο ώστε να, να δώσει το, το, το σήμα και το μήνυμα, τόσο ώστε να γίνει μια έρευνα για, για την υπόθεση των ευρωομολόγων και ιδίω να δούμε υπό ποιε συνθήκε ε, μια τέτοια κίνηση, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορέσει να ωφελήσει όλα τα συμμετέχοντα κράτη, αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Έχετε αντιρρήσει. Όχι φέτο σε ψηφοφορία τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Η τροπολογία 2 κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Δε, κλείνει η ψηφοφορία εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράφος 19 μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 20. Πάλι μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σε κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα. Όχι, δεν είναι ονομαστική κλίση. Το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G. Σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Check, check. στο δεύτερο τμήμα, μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ναι, θα έπρεπε να σηκώσετε τα χέρια σας. Λοιπόν, το σύνολο της πρότασης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται συγχαρητήρια στους συζητητές. Ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία των, ψηφισ... έξι ψηφισμάτων για την κατάσταση στην ακτή Ελεφαντοστού. Καταρχήν το κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων, δεν υπάρχουν τροπολογίες, θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος, κοινής πρώτας ψηφιπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τα τέσσερα ψηφίσματα για την ευζοία των οτόκων ορνήθων. Έξι πολιτικές ομάδες έχουν προτείνει ψηφίσματα. Τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. Όχι, δεν έχει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η 1 έχει από... Τροπολογία 5, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πράγμα σε σε τμήματα Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές από εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τσέκα. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία Επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 8 σε δύο χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ψηφίσουμε την παράγραφο 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 ψηφιπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 4 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας καλύτερα καλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία La Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Χωριστή ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές ε, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί βλέπω ότι δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, με σκέψη F λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συγχαρητήρια. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά και περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου.